Regarding today's... Καλημέρα σα. Για την ημέρησια διάταξη, κατόπιν αιτήματο του κυρίου Γκαμπού, το 6, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλία και Θαλασσών και το 4, ανταλλαγή απόψεων, για τα προϊόντα φωτισμού. Αυτά τα δύο θα ε, αντιστραφούν. Και για να έχουμε καλύτερη ισορροπία μεταξύ των ψηφοφοριών πρωί και απόγευμα, οι ψηφοφορίε για τα 17 και 23 θα γίνουν το πρωί μετά την ψηφοφορία για τα πλαστικά. Αν δεν έχετε αντιρρήσει, μπορούμε να εγκρίνουμε την ημέρα διάταξη με αυτέ τι τροποποίησει. Λοιπόν, στο φάκελό σα θα δείτε τι εκθέσει των αποστολών τη ΕΝΒΗ ε, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος στην Κοπενχάγη 17-18 Σεπτεμβρίου και επίσης ε, στο φόρουμ πολιτικό φόρουμ ψηλού για την ε, βιώσιμη ανάπτυξη στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη στις 16 έως 18 Ιουλίου. Αυτή η αποστολή ήταν κοινή αποστολή με την ΤΕΒΕ. Επίσης, στις 27 Νοεμβρίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα φιλοξενήσει μία υψηλού επίπεδου συνδιάσκεψη με τίτλο η έρευνα και η καινοτομία στην καθημερινή μας ζωή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η βελτίωση της καθημερινότητας των Ευρωπαίων μέσω έρευνας και καινοτομίας, ε, ιστορίες επιτυχίας. Ε, θα γίνει εδώ αυτή η διάσκεψη στο ημικύκλιο, στις Βρυξέλλες. Έχουμε πρόοδους στην ιατρική, καθαρότερη ενέργεια, μηχανολογικά έργα και σε πολλούς άλλους τομείς ε, η έρευνα που χρηματοδοτείται από την Ένωση παίζει ρόλο κλειδί για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Αυτή η διάσκεψη θα είναι μια ευκαιρία να επιδείξουμε τα αποτελέσματα που έχουμε ήδη επιτύχει, αλλά επίση και μια δυνατότητα για αυτού που διαμορφώνουν την πολιτική να ανταλλάξουν απόψει και να προτείνουν νέε ιδέε για την έρευνα και την καινοτομία στην Ένωση με του ενδιαφερομένου, του πολίτε, καθώ και εκπροσώπου των ε, θεσμών τη Ένωση, τα κράτη-μέλη, τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα. Ο πρόεδρο Ταγιάννη και ο επίτροπο Μίδα θα είναι οι κοινοί οι δύο διοργανωτέ, όπου θα ζητηθούν και θέματα ένβη και τα μέλη, και, δηλαδή θέματα ΕΝΒΗ και τα μέλη της ΕΝΒΗ θα παίξουν κύριο ρόλο. Όλη η πληροφόρηση για αυτή τη διάσκεψη και η σελίδα για την εγγραφή είναι στο site του Κοινοβουλίου και θα σταλεί η πληροφόρηση αυτή και στα μέλη μας. Λοιπόν, για σήμερα έχουμε διαρμηνία σε 20 γλώσσες και ως συνήθως μπορείτε να δείτε τη συνεδρίαση στην ε, εφαρμογή e-meeting και η συνεδρίαση μεταδίδεται ζωντανά στο διαδίκτυο. Τώρα, ο μηχανισμός ε, κοινωνικής, ε, πολιτικής προστασίας της Ένωσης. Ο δεύτερος άτυπος τριμερής διάλογος έγινε τη Δευτέρα το απόγευμα στο Κοινοβούλιο. Ξεκινήσαμε μια συζήτηση για θέματα προϋπολογισμού. Είναι σαφές ότι το χάσμα μεταξύ των απόψεων του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου είναι πολύ ευρύ είναι δύσκολο να γεβηρωθεί σε αυτή τη φάση. Ιδιαίτερα λόγω στη θέση του Συμβουλίου που προβλέπει ότι όλοι οι αναγκαίοι πόροι για αυτό το νέο μηχανισμό θα πρέπει να προκύψουν μόνο μέσω ε, μεταφορά πόρων. Η ανταλλαγή συνεχίστηκε με μια συζήτηση για το θέμα τη πρόληψη και το επίπεδο πληροφόρηση που θα πρέπει να ε, ανταλλάσσεται μεταξύ των κρατών μελών και τη Ένωση. Στην πρότασή του, το Συμβούλιο προβλέπει μια, έναν αυτοματισμό μεταξύ ε, διαφόρων ε, επαναλαμβανομένων ε, πυροδοτήσεων και του μηχανισμού επίβλεψης που ε, θα ξεκινάει από την Κομισιόν. Ε, είναι φανερό ότι το Κοινοβούλιο έχει εντελώς αντίθετη άποψη και έχουμε βαριές, σοβαρές μάλλον διαφορές και για τον κανονισμό Rescue δηλαδή πώς θα δημιουργηθεί το σύστημα και αν έχει όντως γνήσια προστιθέμενη αξία. Η Προεδρία θέλει να επιτύχει μια συμφωνία αλλά αντίστροφα από το κοινοβούλιο που έχει κάνει συμβαστικέ προτάσει, δεν έχει κάνει καμία ουσιώδη πρόταση που να αποκλίνει από την αρχική, της, αρχική του στάση, αρχική της τη της Επόμενη άτυπη διαδικασία τριμερούς διαλόγου θα γίνει αρχές Νοεμβρίου. Λοιπόν, πάμε τώρα στο 6 λοιπόν, αυτό που ήταν προηγουμένω. 6 και τώρα γίνεται 4. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θαλασσών και Αλίας. Έχουμε ένα σχέδιο γνωμοδότησης. Ο συγητής είναι ο κύριος Γκάμπους. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Στις 12 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε τη νέα της νομοθετική πρόταση για το Ταμείο Θάλασσας και Αλίας για την περίοδο 2021-27. Όπως ξέρετε, στόχος του Ταμείου αυτού είναι να χρηματοδοτήσει τον προϋπολογισμό της Ένωσης για να στηρίξει την κοινή ελληνική πολιτική, την ναυτιλιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διεθνείς δεσμεύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης στα θέματα διακυβέρνησης των ωκεανών στα πλαίσια του θεματολογίου του 2030 για την βιώσιμη ανάπτυξη. Ως συντάκτης γνωμοδότησης, ε, μάλλον εισηγητής, ε, ευχαριστώ την Επιτροπή μας γιατί θεωρώ ότι η ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι μια πολύ καλή αφετηρία για να καταλήξουμε στην καλύτερη δυνατή συμφωνία. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ισχύ, τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο του Ταμείου, επικεντρώνεται στην προστασία των θαλάσσιων ενδιατημάτων και ε, προτείνει 30% συμβολή συνεισφορά στον προπολογισμό για το μετριασμό των κλιματικών αλλαγών και την προσαρμογή σε αυτή με βάση τη Συμφωνία των Παρισίων. Ευχαριστώ επίσης ε, τις ε, ε, προσπάθειες να ληφθεί υπόψη η περιβαλλοντική βιωσιμότητα και η φορεία, κάτι που με διευκολύνει. Η πρότασή μου απαρτίζεται από τρεις βασικούς πυλώτες, πυλώνες. την συμφόρηση, της, την απαγόρευση αλίας και κυρίως την λήψη υπόψη των περιβαλλοντικών κοινωνικών και κοινωνικο-οικονομικών συνεπειών. Και έχω καταθέσει διάφορες τροπολογίες σχετικά πολύ σημαντικό είναι το θέμα της ε, συμφόρησης. Στην Καταλωνία, στην Καταλωνία έχουμε τέτοιες εμπειρίες με τη συμμετοχή όλων των ε, εμπλεκομένων, δημόσιες αρχές, ε, αλληλείς, επιστήμονες και κοινωνία των πολιτών, μαζί και με μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Και μάλιστα η συνδιαχείριση, συγγνώμη, όχι συμφόρηση, συνδιαχείριση αυτή η διακυβέρνηση στηρίζεται στη λήψη απόψεων με βάση τη γνώση, την ενημέρωση και την αμεσότητα που απαιτείται σε μια ε, οικοσυστημική και βιοοικονομική συνδιαχείριση που ε, τηρεί την αρχή της προφύλαξης. Αυτό το μοντέλο άλλωστε τη συνδιαχείριση αναγνωρίστηκε πρόσφατα από τη ΦΑΟ ω ακολουθητέο μοντέλο για την ελευτική διαχείριση. Και είναι πολύ σημαντική αυτή η αναγνώριση. Αυτό το μοντέλο της συνδιαχείρισης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει μηχανισμούς ώστε να μας επιτρέπει να προσαρμοστούμε στη μεταβαλλόμενη πραγματικότητα με μια προσαρμοστική συνδιαχείριση και επίση το νέο ταμείο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη αυτούς τους νέους μηχανισμούς διαχείρισης των δραστηριοτήτων της ε, επαγγελματικής αλίας, του ψαρέματος αναψυχής και της ε, υδατοκαλλιέργειας με τη συμμετοχή των εμπλεκομένων και την ε, σταδιακή και προσαρμοστική διαχείριση και με μια συνεχή αναθεώρηση ε, και επικαιροποίηση της ενημέρωσης με βάση τις επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις και με ευρεία αποδοχή των εμπλεκομένων λαμβάνονται οι αποφάσεις που επιτρέπουν την εξασφάλιση μιας βιολογικής, οικονομικής και κοινωνικής βιωσιμότητας των τομέων τη επαγγελματική αλίας, τη υδατοκαλλιέργεια και τη αλίας αναψυχή. Επίση, προσωρινό χαρακτήρα τη απαγόρευση τη Για να προσαρμοστεί η αλία στην κατάσταση των αποθεμάτων, θα πρέπει να διατηρηθεί η δυνατότητα ε, παραλυσμού των, των απαγορεύσεων αλίες με βάση βιολογικά κριτήρια στα πλαίσια των αλληλευτικών σχεδίων όπως προβλέπουν οι κανονισμοί. Είναι σημαντικό να κατοχυρώσουμε την αρχή της ανα, αναλογικότητας μεταξύ του διαφυγόντος κέρδους λόγω της εφαρμογής αυτού του περιορισμού της ε, αλληλευτικής προσπάθειας και των αποζημιώσεων. Η αποζημίωση θα πρέπει να είναι σταδιακή ανάλογα με την περίοδο της απαγόρευση αλίας. Επίσης, ε, η διακοπή της ελευτικής προσπάθειας στα πλαίσια του Ταμείου δεν πρέπει να έχουν έκτακτο χαρακτήρα, γιατί ιδιαίτερα ε, κατά την αναπαραγωγή των ειδών που είναι, έχουν κυκλικό χαρακτήρα, είναι επαναλαμβανόμενες αυτές ε, οι διακοπές ελευτικές προσπάθειες Οπότε προσαρμοζόμαστε στην κατάσταση των εχθιαποθεμάτων, λαμβάνοντα υπόψη το, τη διαφύλαξη των θέσεων απασχόληση στο κλάδο. Επίσης, παράκτη αλεία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχειρηματολογεί ότι η παράκτη αεραστεχνική αλεία αντιπροσωπεύει αντιπροσωπεύει το 75% του ευρωπαϊκού ελευτικού στόλου και τις μισέ θέσει απασχόλησης του ελευτικού κλάδου. Γι' αυτό το λόγο θέλει το Ταμείο αλίας να προσαρμοστεί σε αυτό τον αλληλευτικό στόλο, καλύπτοντα ε, όσο περισσότερο μεγαλύτερο τμήμα του γίνεται. Βέβαια, αυτή η επιχειρηματολογία και η διαπροσωπευτικότητα που λαμβάνει υπόψη το μέγεθο των σκαφών και τα είδη, τα, τα είδη των αληφτικών εργαλείων δεν αντιπροσωπεύει όλα τα είδη ε, των σκαφών και των εργαλείων και μερικέ φορέ ε, καλύπτει μόνο το μισό του Ευρωπαϊκού Αλληλευτικού Στόλου, αποκλείοντας μερικές φορές το 83% του αλληλευτικού προϊόντος και άρα θα τρόφιμα και το 90% του οικονομικού βάρους του κλάδου για μερικά αλλιευτικά είδη. Κάτι που συνιστά διάκριση βάρος πολλών ε, αλλιευτικών περιοχών. Γι' αυτό θα πρέπει να συνδέσουμε την έννοια της παράκτησης αλλίας με ε, τα εδάφη, με την τόπια παραγωγή και την στενή σχέση των ελευτικών κοινοτήτων με τον τοπικό πληθυσμό. Επίσης, ε, λαμβάνουμε υπόψη την προστιθέμενη αξία των οπών ακατέργαστων ελευτικών προϊόντων. Θέλουμε επίσης να εξασφαλίσουμε την ε, βιωσιμότητα των λιαυτικών, ε, των ήχθη αποθεμάτων, συγγνώμη, γιατί χωρίς ψάρια φυσικά δεν έχουμε λιαυτική προσπάθεια. Χωρίς αλία δεν έχουμε αλής και χωρίς αλής αφανίζονται χιλιάδες θέσεις, άμεσες και άμεσες θέσεις εργασίας, επηρεάζοντας άμεσα τις τοπικές κοινότητες που εξαρτώνται από την αλεία. Εξού και η ανάγκη να συμπεριλάβουμε τη συνδιαχείριση με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων. Δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω κυρία Πρόεδρε και ελπίζω να συνεργαστούμε με τους και οδησηγητές για να καταλήξουμε σε μια ε, έκθεση με την ευρύτερη δυνατή συνένεση για να εξασφαλίσουμε και τη βιωσιμότητα της τοπικής οικονομίας αλλά και τις θέσεις απασχόλησης στον αλληλευτικό κλάδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Γκαμπούς. Και τώρα να στραφώ στους κοιόδους εξηγητές. Ο πρώτος είναι ο κύριος Τανασέσκου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη σκληρή του δουλειά στην έκθεση αυτή Εκτιμούμε τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επεξεργαστεί την πρόταση αυτή κανονισμού για Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλίας για τη νέα περίοδο 2021-2027 και όπως ξέρετε η πρόταση αυτή σκοπό έχει να υποστηρίξει μέχρι τώρα πρόοδους, την πολιτική αλλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ε, διαχείριση των ωκεανών παγκοσμίω. Καλωσορίζουμε και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να υπάρξει συνέχεια απλούστευση, ε, ευελιξία, ιδίως στη σύνταξη των εθνικών προγραμμάτων με την απαιτούμενη απλούστευση και την ευθυγράμμιση με άλλα ταμεία και κονδύλια. Με την άμεση διαχείριση το νέο Ταμείο για την Αλία και τα θέματα της θάλασσας θα επιτρέψει να υπάρξουν σχέσεις συνεργασίες με άλλα προγράμματα και χρηματοδοτήσεις. Θέλουμε τα αποτελέσματα του Ταμείου να είναι ε, πιο ε, εύληπτα από την περίοδο 2014-2020. Βεβαίω για τον τομέα τη αλεία και τη υδατοκαλλιέργεια δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με 5% μείωση στην, στον προπολογισμό του νέου ταμείου σε σχέση με τον τρέχοντα προπολογισμό. Επίση, οι επενδύσει στην υδατοκαλλιέργεια και την επεξεργασία θα χρηματοδοτηθούν από νέα ε, μέσα, τα οποία θα βασίζονται σε προσωρινό κανονισμό. Όπω ξέρετε, όμω η αλεία και η υδατοκαλλιέργεια έχουν να κάνουν με την επιστηστική ασφάλεια και την ε, διατροφή. Γι' αυτό θα πρέπει το Ταμείο να ε, επιτρέψει να αναπτυχθεί η υδατοκαλλιέργεια. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, θεωρούμε ότι οι επενδύσει στην παραγωγή τη υδατοκαλλιέργεια θα πρέπει να λάβουν την ίδια προκοδότηση με το παρελθόν. Γι' αυτό θα συμφωνήσουμε ότι η χρηματοδότηση είναι σημαντική για την ε, διατήρηση των ε, βιολογικών μας πόρων, την επιστημιστική ασφάλεια, την ε, βιώσιμη οικολογική οικονομία και για την υγεία, την ασφάλεια, την προστασία και την βιώσιμη διαχείριση των ωκεανών. Ευχαριστώ. Thank you. Now, Meissner. Ευχαριστούμε, κυρία Μάισνερ. Er Ευχαριστώ τον εισηγητή είπε πολλά από αυτά που θα ήθελα και εγώ να πω και που θεωρώ σωστά. Από το 2009 ασχολούμαι με την ολοκληρωμένη αλληλευτική πολιτική που είναι από το 2017 μια ευρωπαϊκή πολιτική και θεωρώ ότι είναι απόλυτα σημαντική γιατί οι ωκεανοί παίζουν μεγάλο ρόλο και το βασικό είναι να μην ασχολούμεθα μόνο με την αλία και τις ηχθειοκαλλιέργειες και με όλα, αλλά και με όλα τα άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τη θάλασσα. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό βήμα το ότι διευρύνθηκε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλίας και έγινε Ταμείο Θαλασσών και Αλίας από το 2010. Και ένα μικρό τμήμα των πιστώσεών του ε, στην αρχή χρησιμοποιήθηκε ήδη από την αρχή για την ε, ολοκληρωμένη πολιτική των θαλασσών. Αξιοποιήθηκαν στην αρχή πόροι για την μεταρρύθμιση της πολιτικής αλίας. Ε, είναι σωστό. Πρέπει να κάνουμε πολλά για να υπάρχει βιώσιμη ανάπτυξη της αλίας. Ε, ήταν, ε, τώρα έχουμε 647 για την ε, αλληλευτική πολιτική και άλλα 300 για θέματα που δεν έχουν να κάνουν απευθείας με την αλληλεία. Είναι μικρό ποσό, αλλά παρόλα αυτά είναι μεγάλη επιτυχία γιατί οι πόροι αυτοί συνέβαλαν στην εφαρμογή Τη πολιτική που θα οδηγήσει σε μια μπλε ανάπτυξη, μια βιώσιμη μπλε ανάπτυξη. Αυτό πάντα το θεωρούμε ως μπλε πυλώνα της οικονομίας 2020. Και πιστεύουμε ότι θα δημιουργήσει πάνω από 500 δισεκατομμύρια οικονομικής ανάπτυξης και πάνω από 300.000 θέσεις εργασίας. Πρέπει όμως να καθαρίσουν και οι θάλασσές μας. Και επίσης έχουμε αξιοποιήσει πολλούς πόρους για τη Βαλτική, την, ε, τον Ατλαντικό, την Αδριατική, το Ιόνιο. Αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη ρήπανση στις θάλασσες, την κλιματική αλλαγή. Όλα αυτά χρειάζονται συγκεκριμένε δράσεις από πλευρά της Ένωσης. Σε συνδυασμό βέβαια με το παγκόσμιο θέμα θα ήταν σημαντικό να ε, αναφέρουμε και την ε, διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών. Αυτό έχει αρχίσει να απασχολεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλουμε να είμαστε υπόδειγμα ολόκληρο τον κόσμο. Και αυτά που έχουμε επιτύχει ήδη με την ολοκληρωμένη πολιτική θαλασσών πρέπει να τα διευρύνουμε. Πρέπει λοιπόν ε, να αξιοποιήσουμε τα περισσότερα χρήματα που έχουμε, 829 εκατομμύρια. Δεν είναι και τόσο πολλά, αλλά είναι άλλο ένα βήμα πρόοδου. Και ε, βεβαίως στη θάλασσα δεν υπάρχουν σύνορα και θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την ε, παράνομη αλληλεία, την μόλυνση με πλαστικά. Γενικά πρέπει να καθαρίσουμε τους ωκεανούς, να τους διατηρήσουμε καθαρούς. Και ιδιαίτερα τι ευρωπαϊκέ ακτέ για να έχουμε μια βιώσιμη μπλε ανάπτυξη. Γι' αυτό χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα. Οπότε είναι πολύ καλή αυτή η πρόταση. Χαίρομαι ε, για την περαιτέρω συνεργασία με τον εισηγητή και του περαιτέρω σκιώδη. Ευχαριστώ. Και τώρα η κυρία Έγκστρο. Όχι, δεν θέλει το λόγο. Ωραία. Θέλει κανένα άλλο το λόγο. Όχι. Η κυρία Ζήτοφ από την Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον εισηγητή για αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης, καθώς και όλους ε, τους άλλους που παρενέβησαν και τους οποίους άκουσα πολύ προσεκτικά. Λοιπόν, κάποια σχόλια για την απλούστευση. με την απλούστευση θα μπορούμε να έχουμε πολλές επιλέξιμες δράσεις. Αυτό προτείνουμε. Δεν θα έχουμε έναν αναλυτικό κατάλογο με πολύ περιοριστικού κανόνες. Αντίθετα, θα έχουμε ένα σαφή κατάλογο με μη επιλέξιμες ενέργειες. Όλα τα άλλα θα μπορούν να στηριχθούν. Έτσι τα κρατημέλη θα έχουν πολύ ευελιξία για να προσαρμόσουν τη στήριξη που δίνουν στις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε κράτους μέλους. Οπότε τα σχήματα κοινή διαχείρισης είναι επιλέξιμα. Δεύτερον, θέλουμε να στουρίξουμε καλύτερα την, τους στόχους της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Αλλά σας υπενθυμίζω ότι το ταμείο αυτό είναι και ταμείο θαλασσών δεν μα ενδιαφέρει μόνο η επίτευξη των στόχων τη κοινή αλληλευτικής πολιτική, αλλά θέλουμε να υπάρξουν βιώσιμε υδατοκαλλιτέργειε, να προστατεύσουμε τα οικοσυστήματα και την βιοποικιλότητα στη θάλασσα, την μπλε οικονομία και τις διεθνείς δεσμεύσει τη Ένωση για τη διακυβέρνηση των ωκεανών. Όπω όλοι γνωρίζετε, η ΚΑΠ, η αλληλευτική πολιτική, βασίζεται σε μια προσέγγιση οικοσυστημάτων, δηλαδή η διαχείριση των ε, αλληλευμάτων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τι άλλε ανθρώπινε δραστηριότητε και να συνάδει με την ε, περιβαλλοντική μα πολιτική και τον νόμο. Κυρίω μα ενδιαφέρει να υπάρχει καλό περιβαλλοντικό καθεστώ στι θάλασσε. Αυτό είναι ο οριζόντιο στόχο, στον οποίο πρέπει να συμβάλλει το Ταμείο αυτό. Οπότε, σα υπενθυμίζω ότι η πρόταση περιλαμβάνει επίση και στούριξη προ την ε, Natura 2000. Και προτείνουμε να στηρίξουμε και την συλλογή ε, γνώσης για τις θάλασσες. Έτσι θα βοηθήσουμε ιδιαίτερα τις οδηγίες για τους βιότοπους για τα πτηνά και επίσης θέλουμε μέσω της απευθείας διαχείρισης να συμβάλλουμε και στην προώθηση καθαρών και υγιών θαλασσών και την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα πλαστικά στην κυκλική οικονομία. Επίσης, για τους στόχους ε, διατήρησης των ειδών της ε, κοινής ελευτικής πολιτικής. Θέλουμε να επιτύχουμε περαιτέρω στόχους με σωστή ε, διαχείριση των, του στόλου και με υποχρέωση να εκφορτώνονται τα αλλιεύματα. Επίσης, με βάση την πείρα μας, γνωρίζουμε ότι ορισμένα μέτρα μπορεί να αξιοποιηθούν ούτω ώστε να υπάρχει υπερβολική, υπερβολικό δυναμικό και να μην αξιοποιούνται κάποια μέτρα μόνο όταν υπάρχουν εξαιρετικές περιπτώσεις κρίσης. Γι' αυτό προτείνουμε οι αποζημιώσεις να περιοριστούν μόνο σε ουσιώδη και απρόβλεπτα γεγονότα που ε, έχουν ως συνέπεια ουσιώδη μείωση του εισοδήματος των αλλιέων. Αυτά προτείνουμε και ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Και τώρα κύριε Καμπούς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι εξαιρετικά λακωνικός. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τα καλά τους λόγια. Να πω ότι συμμερίζομαι, αν δεν το καταλάβατε, ε, την πρόταση για απόρριψη της μείωσης ε, του 5% και γενικώ ε, είμαστε στην ίδια γραμμή πλεύσης ό,τι αφορά τη γαλάζια οικονομία και τη βιώσιμη πρώτα απ' όλα οικονομία. Θεωρώ ότι έχουμε λοιπόν πολλά κοινά σημεία και βάσεις για να δρομολογήσουμε μια αξιόλογη έκθεση και είμαι στη διάθεση όλων των σκιωδών εισηγητών και των λοιπόν συναδέλφων ε, και σας υπόσχομαι ότι στο μέτρο του δυνατού θα συμπεριλάβω ε, τις απόψεις στην έκθεσή μου για να ε, επιδώσουμε στην αρμόδια κατουσίαν επιτροπή ε, μια αξιόλογη γνωμοδότηση. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Οπότε Σήμερα εξετάσαμε την έκθεση. Στις 16 Οκτωβρίου λίγη προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας 19 με 20 Νοεμβρίου, ενώ η αρμόδια κατουσία Επιτροπή, Επιτροπή Αλίας, θα ψηφίσει κατά πάσα πιθανότητα τον Ιανουάριο. Οπότε ολοκληρώνουμε τη συζήτηση αυτού του σημείου. Προσπαθούμε να μάθουμε αν θα έρθει ο εισηγητής στο επόμενο σημείο ή όχι. Γι' αυτό περιμένουμε λίγο. Ευχαριστώ. Περνάμε στο επόμενο σημείο, την έκθεση, την εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης για το ενισχυμένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το ΕΚΤ-ΣΥΝ. Η συγγετής μας είναι ο κύριος Μπουσόη, που έχει και το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και λυπάμαι για την καθυστέρηση. Μου είχαν πει ότι στι 10 προβλεπόταν η εξέταση της γνωμοδότησής μου. Εν πάση περιπτώσει, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Πρόεδρε, στις 30 Μαΐου του 2018 η Επιτροπή παρουσίασε πρόταση κανονισμού για την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και της, του κανονισμού για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ΣΥΝ, ένα μηχανισμό ελαστικό ώστε να αντιμετωπιστούν οι προκλήσει τη ε, ενιαία αγορά. Και ενώ ε, πολλοί συμπολίτε μας βρίσκονται στο, στο χείλος του κοινωνικού αποκλεισμού και με διπλάσιο ε, διψήφιο ποσοστό ανεργία σε πολλές χώρες, νομίζω ότι το είναι έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή. Γιατί θα πρέπει να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί στην παγκόσμια οικονομία, να εξασφαλίσουμε ε, το μέλλον σε επερχόμενες γενιές και να έχουμε κοινωνική ένταξη και υψηλά ποιοτικέ υπηρεσίε, παιδεία και υγεία. Ε, Στόχο του ΕΚΤΣΙΝ ε, είναι να συγχωνεύσει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, την Πρωτοβουλία για τους Νέους, ε, το Ταμείο Αρρωγής στους Απόρους, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία και το, Ταμείο για το Πρόγραμμα για την Υγεία προτείνει με ελαστικό μηχανισμό περαιτέρω απλούστευση του προγραμματισμού των κονδυλίων, προκειμένου να μειωθεί περί τη γραφειοκρατία και να εξασφαλιστεί αποτελεσματικότητα προ όφελο όλων των προϊόντων. Βέβαια, το γεγονό ότι συμπεριλαμβάνει στο ενισχυμένο ΕΚΤ και την υγεία δίνει ένα αρνητικό μήνυμα προς Ευρωπαίους πολίτες, ενώ προσδοκούν αυτή η υγεία να παραμείνει προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρόλο που οι αρμοδιότητε τη Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα υγείας δεν είναι σημαντικέ. Καταρχήν, στην γνωμοδότησή μου λέω ότι με τον αυξανόμενο ευρωσκεπτικισμό και στους καιρούς του Brexit θεωρώ ότι θα πρέπει να διαχωρίσουμε το πρόγραμμα για την υγεία, γιατί η συγχώνευσή του διαψεύδει τι προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών. Με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις του Ευρωβαρομέτρου βλέπουμε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτε πιστεύουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επεμβαίνει περισσότερο σε θέματα υγείας. Γι' αυτό θα ήθελα να διαχωρίσουμε τον άξονα υγεία από το ΕΚΤΣΙΝ και να το κατοχυρώσουμε ως ξεχωριστό πρόγραμμα, το πρόγραμμα της υγείας στο επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ευχαριστώ τους συντονιστές που είναι υπέρ αυτή τη Βέβαια, αν δεν καταστηθεί να το κάτι τέτοιο, ελπίζω να έχουμε και ενισχυμένες αρμοδιότητες για το θέμα της υγείας. Σε ό,τι αφορά την ενδιάμεση αξιολόγηση, έχουν διαπιστωθεί σημαντικά επιτεύγματα μέχρι στιγμής. Για να μην μακρηγορήσω λοιπόν και σας κουράσω, θα ήθελα να επισημάνω τα πιο σημαντικά επιτεύγματα. Καταρχήν έχουμε 24 δίκτυα αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ενισχυμένες ικανότητες για να ελεχθούν κρούσματα, στηρίζουμε τις ανάγκες μεταναστών, ε, ενισχύουμε το θέμα ε, της ανείχνευσης και διάγνωσης ε, καρκίνου, AIDS. Έχουμε δραστηριότητες του δικτύου για τα ιατροτεχνολογικά και την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας, γιατί μόνο μόνο το πρόγραμμα υγείας δεν θα μπορούσε στις παραμεθόριες περιοχές να ανταποκριθεί σε όλες αυτές τις προκλήσεις. Με προβληματίζει όμως η μείωση του προϋπολογισμού. Βέβαια η μείωση δεν είναι σημαντική, αλλά παρόλα αυτά εξακολουθεί να είναι μείωση και η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν μας ικανοποιεί. Βέβαια, η μείωση οφείλεται στην ανακατανομή των διαφόρων προτεραιοτήτων στο επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν θα μπορέσουμε όμως ε, αποτελεσματικά και με μειωμένο προπολογισμό να αντιμετωπίσουμε τις σημαντικές προκλήσεις στην υγεία. Το μήνυμα λοιπόν της μείωσης δεν είναι καλό. Και φυσικά στο μέλλον θα πολλαπλασιαστούν οι προκλήσεις που έχουμε. Καλό, θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε. Και γι' αυτό. Για παράδειγμα, η μικροβιακή αντοχή, που γίνεται όλο και οξύτερο πρόβλημα και είναι επιτακτική ανάγκη να βρούμε κοινέ λύσει για να την αντιμετωπίσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Χωρί κατάλληλο προπολογισμό δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε λοιπόν τι πολλαπλέ ε, ε, υγειονομικέ απειλέ και θα να επικεντρωθούμε στην πρόληψη ε, και στην ανάγκη μείωση των ανισοτήτων σε θέματα υγείας, στηρίζοντας τις υγειονομικές υπηρεσίες και καθιστώντας τις οικονομικά προσιτές. Ε, γι' αυτό έχω και σχετικές τροπολογίες. 2, 12 και 70. Επίσης, 458 ε, εκατομμύρια θα πρέπει να είναι σε τρέχουσες τιμές, ε, όπως λέω στις, κατηγο... στις τροπολογίες 13 και 15. Σε άλλες τροπολογίες προτείνω για, τις επι... για τους επιχειρηματικούς στόχους τα εξής. Καταρχήν καλές ε, κοινωνικές παρεμβάσεις και ε, επενδύσεις στην πρόληψη και στον έγκαιρο διαγνωστικό έλεγχο. Με βάση την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, έχουμε 40% των συμπολιτών μας που έχουν κάποιο είδος ε, αναπηρίες. Χρειαζόμαστε λοιπόν μακροπρόθεσμες ε, προσπάθειες για να μειωθούν οι ανισότητες, ιδιαίτερα στον τομέα της υγείας. Επίσης, η οικονομική κρίση επηρεάζει και την ψυχική υγεία. Θα πρέπει λοιπόν να, φροντίσουμε να περιορίσουμε αυτή την αύξηση των κινδύνων. Στο άρθρο 20, στην τροπολογία 20 προτείνω ένα νέο άρθρο 29α. Είμαι υπέρ ενό διοικητικού συμβουλίου για την υγεία και την εφαρμογή των δράσεων στο σκέλος της υγείας και συντονισμό με τα υπάρχοντα μέσα. Και για να επιταθεί η αποτελεσματικότητα των κοινωτικών δράσεων σε διεθνές επίπεδο, θεωρώ σημαντικό να αναπτύξουμε τη συνεργασία με τους, με τους ε, διεθνείς οργανισμούς ΩΣΑ, Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και ούτω καθεξής. Τροπολογία 21. Επίσης, ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μειώσει του φραγμού στη συμμετοχή κάποιων κρατών μελών ε, στο ΕΚΤΣΙΝ. Μερικέ χώρε μέλη βέβαια δεν είναι και πολύ ενθουσιώδες ε, και δεν θέλουν συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα θέματα αυτά. Επίση, πιστεύω ότι η επιτυχία του τρέχοντο προγράμματο θα ενισχυθούν στο επόμενο ενισχυμένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δει πολύ σημαντική εμπειρογνωμοσύνη για τέτοιου είδου δράσει. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα και περιμένω τα σχόλια των σκιωδών εισηγητών και των υπόλοιπων συναδέλφων. Ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη και πάλι για την καθυστέρηση, γιατί νόμιζα ότι η συζήτηση του δικού μου θέματο θα ξεκινούσε στι 10. Κανένα πρόβλημα, κύριε Μπουσόη, κατανοητό. Ο κύριο Πάλμερ που αντικαθιστά την κυρία Κάντεμπαχ ω κοιόδη. Ευχαριστώ. Η κυρία Κάντεμπαχ λυπάται, δεν μπορεί να είναι μαζί μα σήμερα το πρωί. Πρέπει να προεδρεύσει σε μια συνάντηση σχεδόν τη Άγκρη. Έχω τα βασικά σημεία λοιπόν της παρέμβασή τη θέλει να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής ότι στηρίζει τον εισηγητή στο πρόγραμμα υγείας για το Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ αλλά δεν θέλει να ανήκει εκεί ε, ό,τι αφορά την υγειονομική περίθαλψη, να ανήκει σε ξεχωριστή γραμμή του επόμενου πουδουπού. Και καλό θα ήταν να το δει αυτό και η πρόεδρος της Επιτροπής ως μέλος, μέρος της τακτικής δημοσιονομικής διαδικασίας. Επίσης, η μείωση προκοδότησης του τομέα υγείας είναι απαράδεκτη, είναι προτεραιότητα για την πολιτική μας, οπότε θα πρέπει να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τα θέματα της ε, αντίστασης στα αντιβιωτικά και τη μελέτης για τα φάρμακα με την απαραίτητη χρηματοδότηση και φιλόδοξους στόχους για την υγεία και σχετικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να ενθαρρυνθεί η ανάληψη δράση των κρατών μελών σε αυτό το επίπεδο. Γι' αυτό η κυρία Κατενμπάχ ζητά από την Πρόεδρο αυτό να το θέσει στην διάσκεψη των Πρόεδρων. Διότι ήδη είχε συμπεριληφθεί στην ατζέντα τη συνεδρίαση εκεί, αλλά το αφαίρεσαν την τελευταία στιγμή. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε κύριε Πάλμερ και κυρία Γιάτα Μάκη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Όπως ίσως γνωρίζετε δεν είμαι και θειασότης της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν χώνει τη μύτη της εκεί που δεν τις παίρνουν. Αλλά στον τομέα της υγείας Καλό είναι να υπάρξει εμβάθυνση τη συνεργασία για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, να υπάρχει περισσότερη πρόληψη και πιο ε, σφαιρικό σύστημα υγειονομική περίθαλψη στην Ευρώπη. Διασυνοριακά κιόλα και ιδίω εκεί που υπάρχουν κρούσματα και ασθένειε. Με τα νέα τεχνολογικά μέσα και τη γυρεύση του πληθυσμού, η Ευρώπη έχει ανάγκη να αναθεωρήσει εκ βάθρων τα εθνικά συστήματα υγείας και αυτό είναι και μια ευκαιρία για να δει πώς μπορούν να γίνουν πιο ελαφρά ε, στη διαχείριση και πιο παραγωγικά. Πρέπει να καταβάλουμε φιλόδοξες προσπάθειες στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας και τη χρήση των δεδομένων των ασθενών με τρόπο όμως ε, που να υπάρχει πλήρη προστασία των προσωπικών του δεδομένων στι βάσεις δεδομένων. Η ψηφιοποίηση αλλάζει τα πάντα. Τα πάντα από όσα ε, περνάει. Αυτό αφορά και τον τομέα τη υγεία. Τα προγράμματα υγεία, το πρόγραμμα μάλλον υγεία είναι ένα ιδανικό εργαλείο για να υπάρχει ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Η πρόταση για το κοινωνικό ταμείο επικεντρώνεται σωστά στον όρο synergy, σχέση συνεργασίας και τα ενδεχόμενα ωφέλη. Βεβαίως, ε, η λέξη από μόνη της ακούγεται πολύ ωραία, και χρησιμοποιείται για να ε, πούμε πολλά πράγματα. Ελπίζω να γίνει πράξη όμως, γιατί οι σχέσεις συνεργασίας σε αυτό το επίπεδο, ιδίως στον τομέα της υγείας, μπορεί να βελτιώσει τη ζωή των ανθρώπων παντού. Τα έγγραφα που έχουμε ως τώρα για τον προπολογισμό της υγείας καταστούν σαφές ότι η υγεία θα στηριχθεί και από άλλα εργαλεία και μέσα του προπολογισμού, όπως το InvestEU, τα περιφερειακά και διευθυντικά ταμεία και τον ορίζοντα ε, για την Ευρώπη. Όμως θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι λίγο πιο ε, ακριβής ως προς τις συγκεκριμένες συμβολές προς την υγεία από τα συγκεκριμένα αυτά μέσα σε αριθμητικά στοιχεία. Ευχαριστώ για τη συνεργασία των συζητή και περιμένω τα αποτελέσματα των επόμενων συζητήσεών μας. Ευχαριστώ. Thank you very much, Madam Ευχαριστούμε κυρία Κονέτσινα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σπανίως συμφωνώ με συνάδελφο του ΕΛΚ, αλλά εδώ πρέπει να πω ότι δεν έχω ενδιασμούς και δεν έχω και επιφυλάξει για την έκθεση. Μεγάλο μέρο των Ευρωπαίων πολιτών θέλουν η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει περισσότερη δράση στο τομέα τη υγεία. Όμω το τρέχον ε, πρόγραμμα για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο πάει στην αντίθετη κατεύθυνση. Ανησυχώ. Διότι το πρόγραμμα για την υγεία θα πρέπει τώρα να ενταχθεί στο ESF-SYN Θέλουμε να δημιουργήσουμε σχέσεις συνεργασίας μεταξύ της ε, διάστασης των κοινωνικών υποθέσεων και της ε, υγείας. Θετική η προσέγγιση αυτή. Όμως η ίδια η συμπερίληψη της υγείας στο κοινωνικό ταμείο είναι ανησυχητική. Υπάρχουν φήμες ότι στην επόμενη θητεία δεν θα έχουμε και επίτροπο υπεύθυνο για την υγεία και ότι ίσως η Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ να χαθεί ε, μετά την επόμενη θητεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, και αυτό σε μια στιγμή όπου οι Ευρωπαίοι περιμένουν πολύ ενεργότερη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της υγείας. Επίσης υπάρχει και μείωση στον προπολογισμό 8%, κάτι που δεν, είναι δικαιολογη... δεν δικαιολογείται και είναι και παράδεκτο. Επίσης, το ESF θα ε, έχει την πίεση να κάνει περισσότερα με λιγότερα μέσα. Η υγεία δεν είναι μόνο η υγεία του σώματος, αλλά και η ψυχολογική υγεία. Εδώ λοιπόν ε, αποδέχομαι θετικά την πρωτοβουλία του εισηγητή να σχολιάσει και το θέμα αυτό. Όμως, με τα υπάρχοντα μέσα δεν μπορούμε να καλύψουμε όλες τις απειλές που αντιμετωπίζονται. Τώρα που θα υπάρξει μείωση του προπολογισμού. Θα πρέπει λοιπόν ο προπολογισμό να ενισχυθεί, τα προγράμματα για την υγεία να προποδοτηθούν με περισσότερα μέσα και όχι να υπάρξουν περικοπέ. Το Συμβούλιο στο Πολιτέ Δημοσιονομικό Πλαίσιο ε, θα πρέπει να κοιτάξει να βάλει τα προγράμματα της υγείας στο ίδιο επίπεδο τουλάχιστον με το τρέχον. Είναι, το ελάχιστο από το οποίο μπορούμε να ξεκινήσουμε για να παραμείνουμε στην τωρινή κατάσταση που ούτως ή άλλως δεν είναι απόλυτα ικανοποιητική. Θα πρέπει να επιτρέψουμε στους ασθενείς και τις ενώσεις των ασθενών να έχουν λόγο στην όλη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Εδώ συμφωνώ με τον εισηγητή. Είναι σημαντική η διάσταση αυτή στην εκθεσή του και περιμένω τις επόμενες συναντήσεις μας για να συνεννοηθούμε καλύτερα και μαζί του. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκροστέτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με συγχωρείτε για την καθυστέρηση, αλλά ήμουν απασχολημένη σε άλλη συνεδρίαση. Χαίρομαι όμω πολύ που έφτασα εγκαίρω, διότι μπορώ να παρέμβω και να υποστηρίξω τον συνάδελφο Μπουσόη. Έχει κάνει περίφημη δουλειά. Η έκθεσή του είναι τέλεια. Τέλεια από τη δική μου τη σκοπιά δεν προσπάθησε να αποφύγει τους κοπέλους και αυτά που μας ενοχλούν αβολα, γιατί εδώ χρειάζεται τόλμη. Η προοπτική που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμπεριληφθεί η υγεία στο κοινωνικό ταμείο ΣΥΝ, είναι πραγματικά ε, μείζονο σημασία πρόβλημα. Διότι θα κουκουλώσουμε την υγεία σε ένα ευρύτερο σύνολο ει βάρο τη προβολή του και τη αποτελεσματικότητά του. Αυτό είναι εντελώ απαράδεκτο. Όλες ε, οι έρευνες δείχνουν ότι η υγεία είναι σοβαρότατη ανησυχία για τους πολίτες μας και μάλιστα κάτι που τους απασχολεί τόσο πολύ που αλλιώς δεν θα πιστούν για την προστεθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο έτσι θα πιστούν. Ε, Πώ θα του πείσουμε να πάνε να ψηφίσουν στι επόμενε ευρωεκλογέ, Είναι ένα τομέα όπου οι συμπολίτε Θέλουν η Ευρώπη να κάνει πολύ περισσότερα. Το πρόγραμμα υγεία πρέπει να είναι πρόγραμμα που να είναι εντελώ προβεβλημένο, διακριτό και ξεχωριστό στο επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Μιλώ για την Ευρώπη που θα πρέπει να έχει προσθεθέμενη αξία στα υγειονομικά. Εάν ακολουθήσουμε την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ουσιαστικά όλη την ισχύ τη ευρωπαϊκή υγεία θα τη διαλύσουμε. Για ποιο λόγο να ενσωματωθεί με τη συμπερίληψη των μεταναστών, με την απασχόληση των νέων, τι δουλειά έχει. Αντιθέτω, θα έπρεπε το πρόγραμμα υγεία να προβάλλεται και μάλιστα με καμάρι ω ένα ξεχωριστό κομμάτι του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου και του προπολογισμού. Όπω είπε και ο εισηγητή μα, η μείωση των χρηματοδοτήσεων για την υγεία είναι άλλο ένα πρόβλημα. Είναι τελείω ακατανόητε. Οι προκλήσει τι οποίε πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη στην υγεία ολοένα αυξάνονται. Οι προπολογισμοί τη υγεία στα εθνικά κράτη-μέλη ε, γνωρίζουν περικοπέ ενώ έχουμε συνεχώς διακοπές στην παροχή φαρμάκων. Δηλαδή, τα φάρμακα κρυβαίνουν, η έρευνα που επικεντρώνεται σε θεραπευτικές αγωγές που είναι όλο και πιο περίπλοκες. Ο πληθυσμός των ασθενών ε, είναι κατακαιρματισμένος. Οι ε, επιδημίες και οι νόσοι δεν γνωρίζουν σύνορα. Ο πληθυσμός είναι κινητικότερος και η αγορά είναι ενιαία. Το ίδιο και με τα ιατρικά ε, εργαλεία, τα ιατροτεχνικά. Εδώ λοιπόν, ακόμη και το ιατρικό προσωπικό πολλές φορές δουλεύει στο εξωτερικό Όλα τα στοιχεία και τα ηλεκτρονικά δεδομένα των ασθενών δείχνουν ότι πρέπει να έχουν ξεχωριστεί και ιδιαίτερα προβεβλημένη θέση τα προγράμματα υγείας στις πολιτικές μας. Όλα μας καλούν να ανεβάσουμε ταχύτητα για τη συνεργασία μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί εδώ να τραβάει το φρένο για τα προγράμματα υγείας και το ζω κάθε φορά σε κάθε τέλος θητείας. Όποτε πρέπει να σκεφτούμε το μέλλον, προσπαθούμε να πνίξουμε την ευρωπαϊκή πολιτική Υγεία. Ευτυχώ κάθε φορά η πολιτική υγεία σωζόταν. Σωζόταν μόνο και μόνο χάρη στην ε, βούληση τη επιτροπή υγεία και περιβάλλοντο και των βουλευτών που είναι μέλη τη. Ελπίζω ότι για άλλη μια φορά θα είμαστε αρκετά ισχυροί και θα σταθούμε πίσω από τον εισηγητή μα και δίπλα του για να αποφύγουμε να μην ε, συμβεί αυτή η τραγωδία, να χαθεί η ευρωπαϊκή πολιτική Υγεία. Ευχαριστώ. Θέλει κανένα να πάρει το λόγο. Οπότε από την Επιτροπή, η κυρία Κρυσάρ. Α, δεν θέλετε το λόγο. Α. Je préfère passer la parole à mon collègue de la, de la... Ίσως καλύτερα ε, ο συνάδελφός μου από την Γενική Διεύθυνση Υγείας. Α, καλημέρα σας. Είμαι ο Στέφαν Σρέκα ε, από τη Γενική Διεύθυνση Υγείας. Ευχαριστώ τον συγητή και τους Κιώδης για τις απόψεις τους. Ακούσαμε πολύ προσεκτικά και η υπότασή μας που εντάσσει τα θέματα υγείας στο esf SIN εστιάζει στα σημεία που ε, απέδειξαν προστεθέμενη αξία στο παρελθόν. Τα αναφέρατε κι εσείς που πήρατε το λόγο. Εμείς τονίζουμε ότι έτσι θα υπάρχει μία, ένας συνδυασμός το να ενταχθεί το πρόγραμμα υγείας στο esf σύν, θα ε, επιτρέψει καλύτερο συνδυασμό με τις κοινωνικές πλευρές των ενεργειών μας. Οι κοινωνικονομικοί παράγοντες ε, παίζουν μεγάλο ρόλο στα θέματα υγείας. Ακόμη και τώρα. Το κλασικό ESF της, της ε, κοινή διαχείρισης ε, έκανε πολλές επενδύσεις ε, στην υγεία. Και θεωρούμε ότι μπορούν να επιτευχθούν πολλοί συνδυασμοί, πολλές σωστές συνεργασίες, Ούτως ώστε μέσω της απευθείας διαχείρισης της ε, Πλευρά υγεία και μέσω της κοινή διαχείριση ε, άλλων τμήματων του Κοινωνικού Ταμείου στο μέλλον θα οδηγήσουν σε καλύτερα αποτελέσματα. Έχουμε ήδη καλή πείρα και νομίζουμε ότι και στο μέλλον θα έχουμε περισσότερη καλή πείρα. Αυτά ευχαριστώ. Λαμβάνω υπόψη τα άλλα σχόλια. Για τον προπολογισμό, ο προπολογισμό του τμήματος υγείας και των διαφόρων άλλων στοιχείων του ΠΔΠ πρέπει να συνεξεταστούν για να καθοριστεί ο συνολικός προπολογισμό. Οπότε δεν μπορώ να κάνω περαιτέρω σχόλια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος. Ο κύριος Μπουσόη. Ευχαριστώ τους συναδέλφους μου για τα καλά τους λόγια, για την πρότασή μου αλλά και γιατί στηρίζουν την ιδέα να υπάρξει ένα χωριστό πρόγραμμα υγείας και για να αυξηθεί ο προϋπολογισμός. Ο κύριος Πάλμερ από πλευράς της κυρίας Κάντενμπαχ βεβαίω είναι μια απόφαση που θα ληφθεί στη διάσκεψη των Πρόεδρων. Άρα πρέπει να πείσουμε τους επικεφαλείς των πολιτικών ομάδων να μας στηρίξουν. Ευχαριστώ την κυρία Γιάτεμάκη που στηρίζει και εκείνη την ιδέα αύξησης του προπολογισμού. Τουλάχιστον στο να ανέβει στο σημερινό επίπεδο. Και επίσης η ψηφιακή υγεία, η ηλεκτρονική υγεία θα παίξει μεγάλο ρόλο, θα βελτιώσει πολύ την αποτελεσματικότητα, την απόδοση των συστημάτων υγείας. Στην κυρία Κανέτσουνα. Την ευχαριστώ για την στήριξή της. Και Έχω υπόψη μου τις φήμες αυτές για την κατάργηση και της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και του Επιτρόπου Υγείας. Τις θεωρώ απλώς ανόητες. Νομίζω ότι και στο μέλλον η Ένωση θα διατηρήσει την κατάσταση. Γιατί το είπατε σαφώς, ε, η υγεία απασχολεί ιδιαίτερα τους συμπολίτες μας. Τα κράτη-μέλη, οι εθνικές κυβερνήσεις, οι περιφερειακές κυβερνήσεις έχουν την κύρια αρμοδιότητα. Αλλά υπάρχει η προσδοκία ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει περισσότερα. Ευχαριστώ ιδιαίτερα την κυρία Γκροστέτ για τη στήριξή της. Βεβαίως προσθέσατε μερικά στοιχεία στα θέματα που έχω θέσει εγώ για την επόμενη περίοδο. Είναι απόλυτα σαφές. Πρέπει να στείλουμε ένα σωστό πολιτικό μήνυμα. Ενώ τώρα στέλνουμε πολύ λάθος πολιτικό μήνυμα με αυτά που προτείνονται με αυτήν την κατάργηση της αυτονομίας του προγράμματος υγείας. Πολλοί πολίτες μπορεί να το θεωρήσουν και δίκαια ότι είναι το πόδι στην πόρτα. Μας λένε ότι δεν θα εξαφανιστεί η πολιτική υγεία, θα μπει στο ESFC, αλλά αν αποδεχθούμε τώρα αυτό, άμα δώσει τάρος σε αυτούς τους ανθρώπους μπορεί να καταλήξουμε να μην έχουμε πολιτική υγείας ε, χωριστή. Ευχαριστώ πολύ. Και φυσικά και η δική σας προσπάθεια αλλά και το κύρος που έχετε στο Κοινοβούλιο μπορούν να μας βοηθήσουν να ε, έχουμε στήριξη στη διάσκεψη των Πρόεδρων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρος. Πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση. Σας ευχαριστώ πολύ για την έκθεσή σα. Θα ψηφίσουμε μάλλον στις 12 Νοεμβρίου στο Στρασβούργο. Προθεσμία για τροπολογίες 17 Οκτωβρίου. Η Επιτροπή Απασχόλησης, που είναι η αρμόδια επί τη ουσία, θα ψηφίσει στις 26 Νοεμβρίου. Να περάσουμε τώρα στο πρώην σημείο 4, που τώρα έχει γίνει 6 ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή για τα προτινόμενα μέτρα για τα προϊόντα φωτισμού στα πλαίσια του οικοσχεδιασμού και της ε, νομοθεσίας για την σήμανση ενέργειας. Πρώτα η Επιτροπή. Ο κύριος Χότσου. Παρακαλώ. Το πολύ δέκα λεπτά παρακαλώ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καλημέρα. Πρώτα απ' όλα για τη γενική σας ενημέρωση. Τώρα έχουμε πατήσει γκάζι με το πακέτο άνω των 10 τέτοιων πρωτοβουλειών για τον οικοσχεδιασμό και τη σήμανση ενέργειας και αν είναι δυνατόν θα προσπαθήσουμε να το εγκρίνουμε για να το λάβετε πριν τα μέσα Μαρτίου. Έχουμε τον κανονισμό για το φωτισμό ή μάλλον τους κανονισμούς για το φωτισμό. Και δεν έχει ακόμη υποβληθεί πρόταση της Επιτροπής γιατί το Σώμα των Επιτρόπων πρέπει να το αποφασίσει. Εμείς ε, ολοκληρώσαμε τις διαβουλεύσεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα είμαστε στον ε, μηχανισμό ανταλλαγής απόψεων. Μετά θα πάμε στον ΠΟΕ και είτε το Δεκέμβρη είτε τον Ιανουάριο θα ψηφίσει η Επιτροπή Ο φωτισμός είναι πάντα σημαντικό τμήμα της εργασίας μας και με τους κανονισμούς για το φωτισμό που έχουμε ήδη εγκρίνει έχουμε μειώσει κατά 80% περίπου την ε, κατανάλωση ενέργειας από το φωτισμό και με τον στόχο 32,5% εξοικονομής μέχρι το 2030 είναι σημαντικό να μην χαλαρώσουμε, να υπάρξουν περαιτέρω μειώσεις κατά το μισό αυτού που έχει απομείνει. Αυτό είναι δυνατό την επόμενη δεκαετία αν πραγματικά περάσουμε σε διοδική, διοδικό φωτισμό με LED. Θα ακούσω τα θέματα που θα θέσετε, αλλά να αναφέρω τρία θέματα σε αυτή τη φάση, που ήδη έχουν αναφερθεί επανειλημμένα με διάφορους ενδιαφερομένους ε, φορείς. Φωτισμός θεάτρων πρώτα απ' όλα, για τους λαμπτήρες ε, στα θέατρα λοιπόν. Υπάρχει μια ε, εξαίρεση, αλλά αξιοποιείται ως παραθυράκι για να πολλούνται προϊόντα για όλους τους καταναλωτές που υποτίθεται ότι χρησιμοποιούνται από τα θέατρα. και είναι πολύ δύσκολο να δούμε πού χρησιμοποιεί ο καθένας από νομική άποψη κάθε λαμπτήρα. Εντάξει, μιλήσαμε με τον κλάδο. Είναι προφανές ότι ο φωτισμός στο θεάτρο είναι διαφορετικός από ότι ο οικιακός. Γι' αυτό στο σχέδιο του κειμένου μας νομίζω ότι έχουμε αντιμετωπίσει τα περισσότερα θέματα που έθεσε ο τομέας του θεάτρου και θα εξακολουθήσουμε. Η πρόταση λοιπόν, μάλλον, θα εξαιρεί 80% των ε, λαμπτήρων που χρησιμοποιούνται τώρα στα θέατρα, αλλά όχι με βάση την ε, χρήση, αλλά με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά που είναι πολύ πιο ελέγξιμα. Το 20% χρησιμοποιούνται λιγότερο. Είναι αυτά τα προϊόντα που κυρίως είναι αντικείμενα κατάχρησης. Αυτά λοιπόν για τα θέατρα. Το δεύτερο θέμα είναι τα T8. Είναι οι λαμπτήρες φθορίου που έχω και εγώ στο γραφείο μου. Όχι μόνο στα γραφεία βέβαια. Περιέχουν υδράργυρο που πρέπει βέβαια να το δούμε. Και η σταδιακή κατάργησή τους θα μας εξοικονομούσαν 2 με 3 τεραουάτ το χρόνο. Είναι περίπου η κατανάλωση της Μάλτας, άρα δεν είναι αμεληταίο. Η πρόταση που έχει τεθεί είναι να εστιάσουμε στη σταδιακή κατάργησή τους, αλλά αναγνωρίζουμε ότι σε ορισμένε περιπτώσει δεν έχουμε εναλλακτικέ λύσει LED. Ε Γι' αυτό το κείμενο περιέχει και εξαιρέσει. Τρίτο θέμα που συζητήθηκε πολύ για τους προηγούμενους κανονισμούς είναι φωτοευαίσθητα άτομα. Από τη μία πλευρά είναι απόλυτα κατανοητή η ανησυχία τι επίπτωση θα έχουν τα CFL, δηλαδή τα συμπαγή ε, φθοριούχα προϊόντα φωτισμού. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραμείνουν στην αγορά κάποια προϊόντα που είναι παλιά ε, παλιάς Θα επιτρέψει λοιπόν η εξαίρεση για τα φωτευέστητα άτομα να χρησιμοποιούν κάποιους λαμπτήρες, αλλά ε, μόνο με βάση ιατρική βεβαίωση. Στη διάθεσή σας για να ακούσω περαιτέρω ε, παρατηρήσεις και να απαντήσω και σε ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Ποιος θέλει το λόγο. Ο κύριος Λίζε. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και τον κύριο Χότσε. Είναι Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για τα μέτρα που ελήφθησαν για να σώσουν, για να ε, κάνουμε εξοικονομήσεις ενέργειας. Ο Επίτροπος Κατάινεν είπε ότι η οδηγία για τον, οικο, για τον οικολογικό σχεδιασμό Μέχρι πέρυσι είχε εξοικονομήσει την ετήσια κατανάλωση της Ιταλίας και θα μπορέσουμε να προσθέσουμε και την κατανάλωση της Σουηδίας με τα επόμενα μέτρα. Όλα αυτά είναι σωστά. Θεωρώ λοιπόν ότι έχουμε ε, υποτιμήσει πόσο δύσκολο είναι να ενημερώσουμε τι κάνουμε και ποιες είναι εναλλακτικές. Και γι' αυτό παρακάλεσα πριν τα επόμενα βήματα που θα ε, λάβει η Κομισιόν και θα πρέπει και εμείς να δούμε αν τα δεχόμαστε ότι πρέπει να συζητάμε και χαίρομαι που το έχουμε στη μέρη σε διάταξη. Έχω μία ερώτηση για αυτούς λαμπτήρες T8. Γιατί προτείνονται σε αυτή την συγκυρία. Και κυρίως αυτό που με ενδιαφέρει, γιατί αν κατάλαβα καλά, έχετε και εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης ε, Περιβάλλοντος. Με βάση άλλη νομοθεσία, την νομοθεσία ΡΟΣ, συζητάμε πολύ περισσότερο να υπάρχει μια απαγόρευση για τα προϊόντα φωτισμού που όλα αυτά που περιέχουν υδράργυρο. Υπάρχουν ίσως λόγοι αλλά αυτό θα περιόριζε ιδιαίτερα την επιλογή των καταναλωτών. Πρέπει να το σκεφτούμε λοιπόν πολύ συγκεκριμένα και να το συζητήσουμε δημοσίως. Όταν αποφασίσαμε να απαγορεύσουμε κάποιους λαμπτήρες, υπήρχαν κάποιες ε, μελέτες κομισιών που έλεγαν ότι ο υδράργυρος στις, ε, ε στους λαμπτήρες αυτούς δεν ε, είναι τόσο σημαντικός, διότι υπόθηκε ότι ο περισσότερος ε, ε, υδράργυρος στο περιβάλλον προέρχεται από την εξόριξη άνθρακα και ότι αν σταματούσαμε μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας να χρησιμοποιούμε άνθρακα τότε ε, καταργείται ο περισσότερο υδράργυρο και άρα η περισσότερη ε, εξοικονόμηση υδραργύρου που γίνεται μέσω των απτήρων δεν είναι τόσο σημαντική. Και επίση μα λένε και ότι και τα λογόνα καταργούνται συνολικά. Θέλω λοιπόν συνολικά την άποψη τη Κομισιόν. Νομίζω ότι και ο κλάδο και οι καταναλωτέ δεν ενδιαφέρονται για το ποια γενική διεύθυνση θα αναλάβει ε, την πρωτοβουλία. Το θέμα είναι γιατί πρέπει να απαγορευτούν κάποιοι λαμπτήρε. Πρέπει να το συζητήσουμε και να ενημερώσουμε σωστά για να μην έχουμε κάθε εξάμεινο κάποια απαγόρευση από κάποια άλλη γενική διεύθυνση. Πρέπει να τα συζητήσουμε από κοινού, να τα δούμε μαζί όλα αυτά. Ελπίζω λοιπόν αυτή η απαγόρευση που σκέφτεται να επιβάλλει η Γενική Διεύθυνση ε, Περιβάλλοντος, εάν δεν έχει αποφασιστεί ακόμη, να αναβληθεί κατά ένα-δύο χρόνια, γιατί νομίζω ότι η αγορά θα το ρυθμίσει. Οι λαμπτήρες ε, LED είναι τόσο ανώτεροι που θα καταργήσουν τα πάντα. Δεύτερον, η ανταλλαξιμότητα. Το Κοινοβούλιο εξέτασε την έκθεση του Ιράν της Επιτροπής ε, Εσωτερικής Αγοράς, όπου απαιτούσαμε θα πρέπει να έχουμε ανταλλάξιμες πηγές φωτισμού. Δηλαδή, όταν πουλάω ε, ένα φωτιστικό και αν μου χαλάσει το LED μετά από ένα χρόνο να μπορώ να βγάλω την πηγή φωτισμού και να βάλω μια άλλη, να την ανταλλάξω. Και μπορεί να μου αρέσει και το χρώμα του φωτισμού και να θέλω να βάλω κάτι άλλο. Αν κατάλαβα καλά, προβλέπει κάτι η Κομισιόν αλλά προβλέπει μόνο την καλύτερη επιτήρηση της αγοράς. Εμάς μας ενδιαφέρει περισσότερο ο καταναλωτής. Πρέπει να υπάρχει αυτή η δυνατότητα ανταλλαξιμότητας. Και γι' αυτό θα ήθελα η Κομισιόν να το δει περισσότερο από την γωνία του καταναλωτή. Φυσικά υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, δεν μπορεί να τα κάνει κανείς όλα, υπάρχουν κάποιες τεχνικές δυνατότητες και περιορισμοί και πρέπει να τους συζητήσουμε. Αλλά επί της αρχής αυτή η ανταλλαξιμότητα πρέπει να εισαχθεί. Γιατί βοηθάει τον καταναλωτή. Δεν πρέπει να σε ενδιαφέρει μόνο από πλευρά ε, επιτήρηση τη αγορά. Αυτή είναι και η απόφαση που έλαβε πέρυσι το Κοινοβούλιο. Και παρακαλώ λοιπόν την Κομισιόν να το επανεξετάσει. Από την άποψη του καταναλωτή και να μας εξηγήσει τι προτάσεις υπάρχουν τώρα. Σε αυτές τις προτάσει ε, που δεν είναι ακόμη από ό,τι κατάλαβα επίσημε, τι περιέχεται. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, ο κύριος Πάλμερ. Σας ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα του φωτισμού στα θέατρα, γιατί αυτό μας το επισημαίνουν πολλοί και στην εκλογική μου περιφέρεια, κυρίως μικρές οργανώσεις, μικρά θέατρα όπως το Lace Market Theater στο Νότιχαμ, που το διαχειρίζονται εθελοντές ε, ε, και ουσιαστικά χρησιμοποιούν, ε, οργανώνουν μικρές εκδηλώσεις. κάποια κονσέρτα και για τέτοιου είδους μικρής εκδηλώσεις θα θέλαμε να μπορούμε να χρησιμοποιούμε τέτοια την εξαίρεση για τα θέατρα φωτισμού και μάλιστα ε, για τα φωτιστικά στα θέατρα μάλλον. Ε, και μάλιστα περιμένουμε με ανυπομονησία μετά την αναγνώριση από τον κλάδο της ανάγκης εξαίρεσης για το φωτισμό στα θέατρα. Περιμένουμε και με διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους να δούμε ε, τι λύση θα προκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Φαίνεται ότι εισακούστηκαν οι ανησυχίε του κλάδου για, το φωτισμό στα θέατρα, αλλά θα ήθελα να ζητήσω διευκρινήσεις για δύο σημεία είπατε ότι 80% των λαμπτήρων που χρησιμοποιούνται ε, στα θέατρα θα εμπίπτουν στην ε, εξαίρεση. Θα είναι μόνιμη αυτή η εξαίρεση ή μήπω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο μέλλον θα αναθεωρήσει αυτή τη θέση. Γιατί οι αίθουσε και οι οργανώσει που χρησιμοποιούν αυτά τα φωτιστικά και αυτούς τους λαμπτήρες ε, πρέπει να κάνουν έναν ε, επιχειρησιακό προγραμματισμό και οικονομικό προγραμματισμό. Πόσο θα διαρκεί η εξαίρεση, τρία-πέντε χρόνια θα είναι μόνιμη. Επίση, το 20% των φωτιστικών, είπατε, θα πρέπει να αντικατασταθούν και στα θέατρα. Ε, οι πιο ειδικευμένε λάμπε, οι πιο συνήθιστες. Ίσως οι πιο δαπανηρές, οι πιο ακριβές για την κατάσταση θα είναι αυτό το 20%. Οπότε θα έχουμε μια δυσανάλογη συνέπεια για τις μικρές αίθουσε σε σχέση με τα πολύ μεγάλα θέατρα ή τα συναυλιακά κέντρα. Οπότε στις διαβουλεύσεις με τους εμπλεκόμενους και με τον κλάδο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκέφτηκε μήπως ε, ε, θα είναι σκόπιμη μια ενιαία προσέγγιση όταν υπάρχουν τόσες δια... ιδιαιτερότητες και τόσες διαφορές μεταξύ ενός μικρού θεάτρου μιας μικρής αίθουσας εκδηλώσεων και ενός ε, τεράστιου κέντρου συναυλιών που έχει χιλιάδες θέσεις ε, θεατές. Άλλο μια αίθουσα με 50% θέσεις και άλλο ένα τεράστιο συναυλιακό κέντρο. Δεν μπορούμε να εφαρμόζουμε την ίδια λύση για τόσο διαφορετικές αίθουσες. Και σίγουρα θα είναι δυσανάλογο το βάρο τη αντικατάσταση των λαπτήρων. Ακόμη και είναι μόνο το 20% οι λαπτήρε που θα χρειαστούν αντικατάσταση. Σε περίπτωση που μιλούμε για μικρή αίθουσα, ακόμη και για μικρό αριθμό αντικατάσταση, το κόστο θα είναι τεράστιο. Μήπω λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να λάβει υπόψη αυτέ τι διαφορέ και να μην εφαρμόσει μια νέα λύση για όλου, ίσω τελικά να θεωρήσει αυτή τη θέση. Γιατί σίγουρα επειδή έχουμε διαφορετικέ αίθουσε και διαφορετικά μεγέθη, ε, ίσως θα πρέπει να λάβει υπόψη πόσο διαφορετικό θα είναι το κόστος της αντικατάστασης των λαπτήρων ανάλογα με το μέγεθος της αίθουσας των εκδηλώσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Όκεν. Ε, δεν είμαι η Δήμα στα θέματα των φωτιστικών, αλλά είναι πολύ σημαντικό, γιατί η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό ήταν πολύ πετυχημένη. Παρόλο που επικρίθηκε για την ανάμειξη της σε τέτοιου είδους θέματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή απέδειξε ότι καλώς είναι πλάκη και πολλοί καταναλωτές είναι ευγνώμονες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ότι πρότεινε αυτή την οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό. Και αντί να κοιτάει κάποιε θετικέ αξιολογήσει για άλλα θέματα, καλό θα ήταν να εγκύπτει σε τέτοιου είδου ζητήματα. Και το διαπιστώνουμε αυτό. Ε, ακόμη χρησιμοποιούμε τις παλιούς λαμπτήρες ε, τα τελευταία 150 χρόνια, την εφεύρεση του Έντισον. Βέβαια, ακούστηκε ότι οι λαμπτήρες LED ε, όταν ε, ε εφευρέθηκαν, κατηγορήθηκαν ότι το λευκό φως ε, είναι πολύ επιβλαβές, ενώ όλοι χρειαζόμαστε πιο θερμό φως στους παλιούς λαμπτήρες. Και όμως τώρα αποδείχθηκε ότι οι λαμπτήρες LED είναι πολύ πιο οικονομικοί. Επίσης θα πρέπει να προστατεύσουμε τα μικρά θέατρα, τις μικρές αίθουσες εκδηλώσεων απέναντι στις μεγάλες, γιατί θα είναι δύσκολο να αντικαταστήσουν ε, λαμπτήρες ε, όταν το έξοδο θα είναι τεράστιο, ειδικά οι μικρές αίθουσες. Βέβαια, από την άλλη, όταν μπορούμε να κάνουμε κάποιε οικονομίε στην ενέργεια, καλό θα είναι να το κάνουμε. Θεωρώ ότι η πρόταση τελικά είναι καλή και ασκεί τι πιέσει εκεί που χρειάζεται. Βέβαια, πολλά είναι τα παραδείγματα και πολλοί μας λένε ότι κάποιε δραστηριότητες θα κλείσουν αν δεν μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν το, τα παλιά μοντέλα λαμπτήρων. Θα πρέπει να βρούμε μια βιώσιμη λύση και για τα μικρά θέατρα και για τις μικρές αίθουσες ε, εκδηλώσεων. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγγύψει και σε αυτό το θέμα. Επίσης, περιμένουμε τις προτάσεις για τον οικολογικό σχεδιασμό. Είναι καλή ιδέα. Περιμένουμε προτάσεις για εύχριστα για τους καταναλωτές προϊόντα. Και φυσικά μία εύκολη εφαρμογή ώστε να αποφευθούν παραθυράκια. Ο καταναλωτής χρειάζεται ένα εργαλείο που θα είναι καλό για το περιβάλλον, αλλά και εύχριστο για τον ίδιο. Περιμένουμε λοιπόν από την Οδηγία για το Οικολογικό Σχεδιασμό ένα μηχανισμό που να λειτουργεί. Πάντω, μέχρι στιγμή οι προτάσει είναι πολύ θετικέ και περιμένουμε το συνολικό πακέτο. Ευχαριστώ. Okay, thank you. Ευχαριστούμε πολύ. Άλλο κανεί από του θέματο, εάν όχι, ο κύριο Χάτσον. Ευχαριστώ και πάλι, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλα τα μέλη της Επιτροπής σας που εξέφρασαν και τη στήριξή τους για το πρόγραμμα συνολικά. Βεβαίω, οι μισέ εξοικονομήσει ενέργεια που πετυχαίνουμε αυτή τη δεκαετία έχουν να κάνουν ε, με την ε, αλλαγή στην επισήμανση τη ενέργεια και τον οικολογικό σχεδιασμό. Και στα σπίτια και στα εργοστάσια, με τι αλλαγέ που έχουν γίνει, γίνονται συνολικά πολλέ οικονομίε. Στον κύριο Λίζε, να πω, όπω και στην κυρία Όκεν, ότι χρειάζεται καλύτερη επικοινωνία, ιδίω όταν αλλάζουμε τι ετικέτε. Μέρο τη νομοθεσία που συμφωνήθηκε πέρσι. Θα συνεργαστούμε με τι εταιρείε, με τα κράτη-μέλη, για να έχουμε την ευκαιρία να εξηγήσουμε και στου καταναλωτέ πώ χρησιμοποιούνται οι νέε επισημάνσει, ιδίω για τα προϊόντα υψηλή προτεραιότητα, πώ μέρο αυτή τη δέσμη μέτρων θα περάσουν πρώτα. Πάλι στον κύριο Λίζε, να πω ότι έχω εδώ συνάδελφο την DJ Envy και έχουμε συνεργαστεί στενά για το πακέτο αυτό και για τις ε, προτάσεις για τα πλυντήρια πιάτων και τα πλυντήρια ρούχων και για όλη την ε, προσπάθεια εξοικονόμησης σε όλο το πακέτο. Τώρα στο γενικότερο θέμα του υδράργυρου στους λαμπτήρες Υπάρχει στην ισχύουσα νομοθεσία ε, η απαγόρευση για τι επιζήμιε ουσίε. Η αναθεώρηση αυτή δεν έχει καταλήξει ούτε στην μια κατεύθυνση ούτε στην άλλη. Και εμεί θα σημειώσουμε τι δικέ σα παρατηρήσει για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και να συζητήσουμε πρωτού καταλήξουμε σε απόφαση και γίνει αλλαγή στην νομοθεσία. Ω προ του φθορίζοντα, τους φθορίζοντες λαπτήρες T8, η αλλαγή που προτείνεται τώρα είναι να δούμε τι στιγμή υπάρχει τώρα ως προς τα LED, τι εναλλακτική υπάρχει τώρα ως προς τα LED και τι οικονομίες μπορούν να γίνουν. Είναι η κλασική προσέγγιση. Δεν πρόκειται για κάτι καινούριο. Ένα παρελκόμενο όφελος θα είναι ότι θα χρησιμοποιούνται πολύ λιγότερο οι λαμπτήρες ετραγύρου. Ο κύριος Λίζε έχει δίκιο που θυμίζει τις συζητήσεις που είχαμε για τον Τζάργυρο τον οποίο αποφύγαμε με τη μειωμένη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, οπότε δεν είχαμε κίνδυνο να υπάρχει η διάχυσή του στο περιβάλλον από τους λαμπτήρες. Θα πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε πώς θα αποφύγουμε περαιτέρω τον κίνδυνο αυτό. Μετά για τις ε, πηγές φωτισμού που θα είναι ανταλλάξιμες, δεν έχουμε πάει τόσο μακριά για την ώρα στα μέτρα μας, τόσο μακριά όσο ζητά ο κύριος Λίζε ή τέλος πάντων η έκθεση που ανέφερε μαζιτά, Επιμένουμε ότι θα πρέπει να είναι δυνατόν για τις αρχές εποπτείας της αγοράς να τεστάρουν, να δοκιμάσουν τους λαμπτήρες που πολλούνται στην αγορά τους για να είναι βέβαιος ότι είναι συμβατές με τις απαιτήσει αλλά αυτό μπορεί να γίνει με δύο διαφορετικού τρόπου βάσει του κειμενικού του πίνακα. Δηλαδή, είτε με την απομάκρυνση και την κατάργηση ενό λαμπτήρα, είτε με το να βεβαιώνονται ότι η συσκευή που περιέχει ο λαμπτήρα μπορεί να δοκιμαστεί. Και αυτό γιατί στι συζητήσει που είχαμε με τι εταιρείε ε, και την, τον όλο βιομηχανικό κλάδο είδαμε ότι θα είναι υψηλότερο το κόστο υψηλότερο το κόστο τη απομάκρυνση από την αγορά ενό ολοκληρωμένου προϊόντο και εδώ είναι και η ευρωπαϊκή προστεθέμενη αξία η ευρωπαϊκή υποστηθέμενη αξία. Διότι αν δεν φύγει η παραγωγή από την Ευρώπη, η δουλειά των Ευρωπαίων σχεδιαστών με τη μεγαλύτερη ευελιξία που τους προσφέρεται, θα μας προσφέρει και οικονομική δυνατότητα. Γι' αυτό δεν θέλουμε να υπάρχει ανταλλαξιμότητα σε όλες τις περιπτώσεις. Στον κύριο Πάλμερ και την κυρία Άουκεν, για το φωτισμό στα μικρά θέατρα και για την ε, διάρκεια. Δεν υπάρχει όριο στη διάρκεια και για τις εξαιρέσεις ε, βέβαια της πρότασης. Για συγκεκριμένες ε, πρίζες και πηγές είναι συγκεκριμένη διάρκεια. Όσα επιτρέπονται θα επιτρέπονται και θα μείνουν στην αγορά. Η ρήτρα αναθεώρησης που υπάρχει στο κείμενο έχει προβλέψει πενταετία μετά τη θέση σε ισχύ. Όμω δεν υπάρχει συγκεκριμένη πρόθεση να αλλάξουν οι, φωτισμοί για το, να, διατάξει για το φωτισμό των θεάτρων εν μεταξύ. Για το 20% δεν ήμουν πολύ σαφή. 20% των κατηγοριών λαμπτήρων, όχι 20% των λαμπτήρων συνολικά, είναι πολύ λιγότερο. Είναι ένα μέρο του ποσοστού για το ίδιο και για το φωτισμό των θεάτρων στα μικρά θέατρα είναι ειδικό ο φωτισμό, είναι ειδικοί οι λαμπτήρε, δεν είναι οι ίδιοι με τι μεγάλε συναυλιακέ εγκαταστάσει. Είναι συγκεκριμένα τα είδη που θα επηρεαστούν στα μικρά θέατρα και πολύ περιορισμένα. Είπα προηγουμένω ότι θα υπάρχει ένα μηχανισμό feedback απόκριση, κάτι που σημαίνει ότι μετά από τέσσερι εβδομάδε από τη θέση ισχύει κάπου τώρα, και μετά τι διαβουλεύσεις που έχουμε κάνει και παρόλα αυτά, παρόλο που είμαστε σε προχωμένο στάδιο τη διαδικασία, εάν υπάρξουν ανησυχίε, θα τις λάβουμε υπόψη. Είμαι βέβαιος ότι όσοι ασχολούνται με το φωτισμό των θεάτρων, οι φωτιστές θα ενημερώσουν. Θα κοιτάξουν το κείμενο ω έχει σε αυτή τη φάση και θα δούμε εμεί τι μπορούμε να κάνουμε από την πλευρά μα. Δύο σχόλια ακόμη ο οικολογικός σχεδιασμός λειτουργεί ω εξή. Δεν υποχρεώνεται κανεί να πετάξει του λαμπτήρε του ή το πλυντήριο του ή την ηλεκτρική του σκούπα. Ε, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να μην υπάρχουν πλέον ε, άχρηστα προϊόντα στην αγορά. Να κρατήσει κανεί ε, ό,τι έχει, αφού το θέλει, μέχρι να σταματήσει να λειτουργεί. Η απέτηση αρχίζει να ισχύει, αλλά δεν υποχρεώνει σε τίποτα. Φυσικά κόστος θα υπάρξει. Αλλά όταν είναι καλή αντικατάσταση με LED, το κόστος ζωής τελικά προσφέρει οικονομία. Θα κρατήσει πολύ περισσότερο η διάρκεια ζωής και θα εξοικονομεί κανείς ενέργεια. Αυτό ισχύει και για τα θέατρα. Η οικονομική εξίσωση έχει να κάνει περισσότερο με το ότι τα θέατρα μπορούν να συνεχίσουν να είναι το ίδιο ωραία όπως είναι και τώρα, αντί να κοιτάξουμε μόνο πώς θα μειώσουμε το κόστος αλλά στις συνεχιζόμενες συνεζητήσεις μας μπορούμε να το δούμε ξανά. Και μια τελευταία παρατήρηση. Αύριο ξέρω ότι κοιτάζετε την αναθεώρηση του προγράμματος LIFE. Έχει προβλεφθεί στην ατζέντα σας. Να ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλη η δουλειά που κάνουμε για την υποστήριξη του οικολογικού συνδυασμού ε, και τη νέα επισήμανση και η δουλειά που κάνουμε για τις βοπτικές αρχές και την υποστήριξη της επιθεωρήσης και ό,τι κάνουμε για το LIFE έχουν όλα να κάνουν με του προβαλλοντικούς μα στόχου. Οι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πρόγραμμα LIFE στην επόμενη περίοδο έχουν να κάνουν και με τη μετάβαση της καθαρής, στην καθαρή ενέργεια. Θα είναι μέρος του προγράμματος LIFE αυτό στο επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Απλώς σας το είπα έτσι ενημερωτικά ως προειδοποίηση. Ε, αυτά και με την Γενική Διεύθυνση Ενέργειας. Να ξέρετε ότι και με, τους συναδέλφους μας που με τον συνάδελφό μας που εργάζεται για τα θέματα αυτά είμαστε στη διάθεσή σας για να απαντήσουμε σε τυχόν ερωτήσεις. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ολοκληρώνουμε τη συζήτηση πριν τις ψηφοφορίες. Οι ψηφοφορίες προβλέπονται στις 11, οπότε αυτή τη στιγμή θα πρέπει να διακόψουμε. Έτσι θα μπορέσετε να συνεχίσετε τα πηγαδάκια σας. Και αν θέλετε με τον κύριο Σενάντερ και την ομάδα του.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 Well, hello everyone. If you want to take your... Χαίρετε. Παρακαλώ καθίστε. Και ε, βγάλετε και τις κάρτες σας. Ψηφοφορίας. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε και δύο άλλα θέματα που ήταν να ψηφίσουμε το απόγευμα. Θα τα ψηφίσουμε τώρα το πρωί. Είναι το 17 και το 23. Σας παρακαλώ, εφόσον έχετε έτοιμες τις ε, κάρτες ψηφοφορίας σας. Κύριε Φαρία, γιατί τα περάσατε το πρωί αυτές τις δύο εκθέσεις. Μπορεί να μας εξηγήσετε παρακαλώ γιατί δεν το μάθαμε. Είναι μια απόφαση που πήραμε τη γραμματεία για να έχουμε περίπου τις ίδιες ψηφοφορίες πρωί και απόγευμα. γιατί είχαμε πολύ περισσότερες το απόγευμα. και έχουμε πολλές ε, τροπολογίες συμβαστικές για τα πλαστικά. Οπότε, πρώτα απ' όλα, να ψηφίσουμε την προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ψηφιακή ε, μεταρρύθμιση του, ε, της αγοράς για τα προϊόντα υγείας. Ε, ηλεκτρονικά άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Να ψηφίσουμε για την προφορική ερώτηση για τις σπάνιες ασθένειες. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Να ψηφίσουμε για μια ερώτηση για προφορική απάντηση για μια Ευρώπη που προστατεύει τον καθαρό αέρα για όλους. Άρχεται. Και πέρας. Και εγκρίνεται. Τώρα να ψηφίσουμε προφορική ερώτηση για την πρωτοβουλία για τους επικονιαστές. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τώρα, να ψηφίσουμε για τη μείωση της επίπτωσης κάποιων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον. Τροπολογία 46. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 11 ένα, συγγνώμη, ε, εγκρίνεται. Τροπολογία 2.30. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2.31. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2.32. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Άγκρη 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 2. Υπέρ κατά αποχές δεκτή 2.43 και 2.44 ήτρε 36 και άκρη 33 ταυτόσιμες υπέρ παρακαλώ κατά αποχές απορρίπτονται 2.42 υπέρ υπέρ λοιπόν κατά αποχές απορρίπτεται Τώρα να ψηφίσουμε τη συμβαστική 5 υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές δεκτή. ...266 και άγγελ 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 267 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Πες 25 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 14 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 10 υπέρ. <clears throat> Κατά αποχές δεκτή. 2.41 υπέρ Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.63 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.76 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Α, έλεγχος. Πέρας. Δεκτή. Ευχαριστώ πολύ. Οι άλλε οι επόμενες δύο καταπίπτουν. Να ψηφίσουμε την 22 υπέρ παρακαλώ. <clears throat> Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Στη σελίδα 10. 2,78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 4α υπέρ κατά αποχές δεκτή. Και ως προσθήκη τώρα να ψηφίσουμε τη συμβαστική 4β υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Μ, έλεγχος. Πέρας. Δεκτή. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 3.54 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Α, είναι ταυτόσιμη με 3.55. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Στη σελίδα 16. Αλία 28, πες 28. Το δεύτερο τμήμα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Άρχεται. Ε, πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Τι κάνει το ECR. Αλλά νομίζω ότι εγκρίνεται. Έλεγχο. Πέρας. Δεκτή. Συμβαστική εννέα. Υπέρ. Κάτα. Αποχές συγκρίνεται Σελίδα 22, συμβαστική 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές Δεκτή. 4,75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έκον 25 και Ήτρε 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 4,76 έχουμε μία κατά τμήματα ψηφοφορία. Το πρώτο τμήμα, ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 4,77 υπέρ. Κατά έλεγχος. Άρχεται. πέρασε, Δεκτή. 4,78 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Έκον 26 και Ήτρε 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 4,80 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Α, έλεγχος. Τις 4,80. Άρχεται. Πέρασε. Δεκτή. Συμβαστική 12 υπέρ κατά Αποχές. Δεκτή. 4,90 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές. Δεκτή Σελίδα 29. 522. Υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος. Πέρας. Απορρίπτεται. Ήτρε 59 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 526 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Πάμε στη σελίδα 37. Τροπολογία. 621. 22, 23, 24. Και μία προφορική τροπολόγηση από τον εισηγητή. Πού την έχετε γραπτή. Επειδή υπάρχει προφορική τροπολόγηση, πρέπει να ρωτήσω εάν υπάρχουν αντιρρήσεις. Όχι. Καλώς. Θα ψηφίσουμε και αυτήν την προφορική τροπολόγηση. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Άγκρι 79 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Σελίδα 44. Άγκρι 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν βλέπω να σηκώνετε τα χέρια σας. Επαναλαμβάνω. Άγκρι 1. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Στη σελίδα 44. Το είπα. Έκον 1 και 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Έκον 2 και Ήτρε 5. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 53 υπέρ κατά αποχές έλεγχος της 53. Τέλος, εγκρίνεται. 54. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεν βλέπω ξεκάθαρο το αποτέλεσμα, ηλεκτρονικός έλεγχος. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ήτρε 2. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Άγκρι 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 55. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, αλία 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ήτρε 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 57. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 58. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 59. Ε, καταπίπτει. 60. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 61 και ήτρε 6. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Απορρίπτονται. 63. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 64 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Έκον 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 66 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αλία 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται άγκρι 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 71. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 71. Άρχεται ψηφοφορία. Αν και νομίζω ότι εγκρίνεται. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται όντως. Αλία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5 και άγκρι 6. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Ήτρε 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 73. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αλία 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Σελίδα 48. Ε, 9. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος. Εγκρίνεται. 91. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 92 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Άγριε 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 104. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αλία 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 13 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 24 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 21 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 12 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 16 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 14 υπέρ. Κατά αποχές το ΕΛΚ υπέρ επανάληψη ψηφοφορίας Ήτρε 14 ποιος είναι υπέρ α εγκρίνεται γιατί απορρίψαμε σχεδόν όλες τις τροπολογίες της Ήτρε και της Ελίας. Άκρη 14. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 115 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 15 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 118 υπέρ. Κατά. «118 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται». 120 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος μάλλον. And close. EPP plus one. Απορρίπτεται. 119, who is in favor. 119. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 15. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Περνάμε στη σελίδα 51. 130 και 8. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Απορρίπτονται. 131. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 141 στην επόμενη σελίδα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 150 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 151 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 152 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Αλία 12. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Αλία 12. Υπέρ πρώτα. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αλία 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εκόν 11. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έκον 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 179 και άγκρι 10 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. Άγκρι 21 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 180 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 22. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. And it's closed. Τέλος ψηφοφορίας. Έχει εγκριθεί τελικά. Mm. Αλία 18. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 25 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 204 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 30, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 217 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 218 και άγκρι 29. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 219. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 220 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 200... 221 την ψηφίσαμε. 221 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 222 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας και εγκρίνεται. Now, now we vote on... Θα ψηφίσουμε τώρα μια γνωμοδότηση για την πρόταση κανονισμού Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για αποκαλύψεις που αφορούν τις βιώσιμες επενδύσεις και την τροποποίηση της οδηγίας 2341 συγγνώμη, του 2016. Αλλά πρέπει να σηκώνετε τα χέρια για να βλέπω το αποτέλεσμα. Τροπολογία πρώτη. Υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχος. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 31 και 32. Υπέρ. Κατά. Με συγχωρείτε. Συγγνώμη. 31 μόνη της. 31 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος, επαλήθευση, 34.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 αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος για το 54. Πέρας. Εγκρίνεται. 55 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 57 υπέρ. Κατά. Υπέρ το ΕΛΚ. Εγκρίνεται. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 60 υπέρ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 Πέρας. Εγκρίνεται. Με μία ψήφο διαφορά. Η 72 δεν ψηφίζεται. 2. Υπέρ. Με κατά αποχές απορρίπτεται. 3. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 4. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, απορρίπτεται, συγγνώμη. 6. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 5. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 14 υπέρ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 28 συγγνώμη υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 30 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονική, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Νομίζω ήταν το τελευταίο για σήμερα το πρωί. Α. Και τώρα, γνωμοδότηση για κοινέ διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο ε, και Θαλάσσιων Υποθέσεων, για το άσυλο και τη μετανάστευση, και ούτω καθεξής. Ξεκινάμε με την τροπολογία 36 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Νομίζω εγκρίνεται, αλλά για να είμαστε βέβαιοι. Εγκρίνεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ. 38 έλεγχος. Πέρας. Απορρίπτεται. Ευχαριστούμε. 39 υπέρ. Κατά έλεγχος. Δεν είναι σαφής ο διαχωρισμός. Εγκρίνεται. 40 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 41 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 42. Έλεγχος. Επαλήθευση. Πέρας, εγκρίνεται. Σαράντα δύο υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 43 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Πέρας. Απορρίπτεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος για την 45. Πέρας. Εγκρίνεται. 46 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 48 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 49 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 50 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 51 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 52 υπέρ, κατά,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 Επτά υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την επτά. Πέρας εγκρίνεται. Εννέα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δέκα υπέρ κατά αποχές δεν βλέπω την άλλη στη μέτρηση. Είναι υπέρ ή κατά. Τότε εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 15 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά έλεγχος για τη 16. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 25 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 27 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 28 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 30 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 31 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 32 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονική αυτή, άρχεται. Και πέρας εγκρίνεται. Ολοκληρώνουμε με τις ψηφοφορίες για σήμερα το πρωί. Σας θυμίζω ότι έχουμε ακόμη μία το πρωί, το απόγευμα, στις 4. Σας ευχαριστώ πολύ.